Για δυόμιση λεπτά έχει τον λόγο η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτός ο συγγραφέα αλλά και ακτιβιστής των ποινών δικαιωμάτων καταδικάζεται σε 11 χρόνια κάθεξη διότι έδωσε μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από ένα χρόνο είχε συλληφθεί μετά από αυτή τη χάρτα δικαιωμάτων που προσυπέραψαν πάνω από 10.000 πολίτες και ζητούσαν τα πιο φυσιολογικά πράγματα για μια δημοκρατική κοινωνία. Το δικαίωμα λόγου, ελεύθερες εκλογές, κράτος δικαίου, η καταδίκη του Λιούσοβο ε, οφείλεται σε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, υπέστη δικαστική δίωξη, κάτι το οποίο όμως είναι κάτι που δεν συμβάζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τις θεμελιώδη ελευθερίες. Θα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωσή του. Συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας περιορίζονται στην οικονομική διάσταση. Οπότε παραμελείται η κακή επιδοσή της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα, η συστηματική τους παραβίαση οι αστυνομικοί έχουν παραδεχτεί ότι ο Σι Σισέγγ που είναι νομικός λαμπρός και αγωνιστής για ανθρώπινα δικαιώματα αγνοείται ενώ κρατείται από τις διοικητικές αρχές και πολλοί φοβούνται ότι έχει πεθάνει παρά το ότι έχει γίνει έκκληση να μην εκτελεστεί διότι είναι Βρετανό πολίτη. Για πολλωστή φορά, από μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνώρισαν οι Κινέζοι τι εκκλήσει τη διεθνή κοινότητα. Επομένω, με όλα αυτά τα δεδομένα, από πού και ω πού ε, η Κίνα θέλει να συμμετάσχει στο Συμβούλιο του ΟΗΕ τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί για να νομιμοποιήσει αυτέ τι λιβερέ τι επιδόσει. Ήδη έχουν ε, διακηρύξει με ένα μακροσκελέ έγγραφο ότι θα ένα πρόγραμμα για αποκατάσταση δικαιωμάτων, το οποίο είναι νεκρό γράμμα βέβαια. Οπότε θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρήσει ότι υποχρεούται να κάτσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του διαλόγου Ένωση Κίνα. Ευχαριστούμε κύριε Βέμπερ και τώρα. Για ένα λεπτό έχει το λόγο κύριο Κέλαμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Κίνα έχει εντυπωσιακή οικονομική πρόοδο όμως εν μέρει αυτό έχει επιτευχθεί με μέσα τα οποία παραβιάζουν πλήρως τις διεθνείς διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίδες ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες θα παρακινούσαν τις κινέζικες αρχές να σεβαστούν τις δημοκρατικές αρχές αγουδίχθηκαν μάταιες. αυτού συνεχίστηκε η καταπίεση και πρέπει να βγάλουμε κάποτε συμπεράσματα. Σήμερα καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την μοίρα του Λιού Σαββάου, ενός λόγιου, ο οποίος είχε υπογράψει την χάρτα του 2008 για την περάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας χάρτας η οποία συνυπεγράφει από πάνω από 10.000 γενναίους και νέους πολίτες, είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του σε 11 χρόνια φυλάκιση. Σήμερα ζητάμε την άμεση και ανεφόρον αποφυλάκησή του και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τις ειρηνικές πράξεις των Κινέζων πολιτών υπέρ της δημοκρατίας και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγματα για τα οποία έχει δεσμευτεί η Κίνα. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλαμ για δύο λεπτά η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ψηφίσματα ε, ε, επί κατεπηγόντων συνήθως είναι δύσκολα πράγματα, γιατί ε, συνήθως αντί να καταδεικνύουν μια ανθρωπιστική κατεπήγουσα κατάσταση, καταδεικνύουν την πολιτική μας αδυναμία. Τα... Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα μέσα διαλόγου και δράξη... δράσης έχουν αποτύχει και αντί να δράσουμε απλώς καταδικάζομαι επανειλημμένα έχουν ε, πολλά ψηφίσματα έχουν περάσει από εδώ αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν αποτέλεσμα ή δεν είχαν αποτέλεσμα το να επανερχόμαστε όμως διαρκώς ε, στην επίθεση δεν σημαίνει ότι κάνουμε λάθος στην πολιτική μας, αλλά ε, σημαίνει ότι έχουμε κάνει λάθος όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος θανατικές εκτελέσεις, ε, ξυλοδαρμοί, ε, παραβιάσεις. Ε, γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Επίσης γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί με τον Λιού Ξαομπό καθώς και επίσης με τον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί σύμβολο της πλατείας Τιενανμένα. Όμως εμείς χρειαζόμαστε ε, την χώρα αυτή. Πρέπει να είναι εταίρος μας ε, για τις πολιτικές εξελίξεις, για την ισορροπία σε όλο τον κόσμο, για τις κλιματικές αλλαγές. Επομένως, ε, για πολιτικούς λόγους πρέπει να βρούμε δρόμο συνεργασίας με τη χώρα αυτή. Για αυτούς τους λόγους αποσύραμε την πολιτική μας υπογραφή από το ψήφισμα. Όμως, θα ψηφίσουμε υπέρ όλων των τροπολογιών ε, που έχουν ε, υποβληθεί για να μην υπάρξει καμία παρανόηση όσον αφορά την πολιτική μας τοποθέτηση. Για δύο μισή λεπτά η κυρία Βερζιά. Η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα με πλούσια ιστορία και με ε, αστήρευτο δυναμικό ανάπτυξης η προσπάθεια που έγιναν την προηγούμενη χρονιά και οι ε, Ολυμπιακοί Αγώνες ε, δεν κατάφεραν ε, να δώσουν την τροπή που περιμέναμε όλοι. Σαν Ευρωπαίοι βουλευτές εμείς θα πρέπει να βροντοφωνάξουμε αυτά τα οποία θεωρούμε άδικα και απαράδεκτα. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα αυτή δεν είναι απαράδεκτα. Ε, και ε, βεβαίως ε, ο Λίου Ξιάομπο γνωρίζομαι ότι κατάφερε να κινητοποιήσει 10.000 ανθρώπους και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους όπως ο Λιου Ξιαομπό και όλους όσους ε, θεωρούνται εγκληματίες ε, γιατί προσπάθησαν απλώς να εκφραστούν ελεύθερα. Όπως ε, είπε και προηγουμένως ένας συνάδελφος, εκτελέστηκε θανατική ποινή όσον αφορά Βρετανό υπήκο, ενώ ενώ επρόκειτο για άτομο που αντιμετώπιζε πνευματικά προβλήματα. Η περίπτωση του Google που ε, παρόλα αυτά ε, είναι ένας ε, operator ο οποίος ε, δεν φημίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά παρόλα αυτά θέλει να προστατεύσει τους χρήστες του. Καταλάβαμε τι γίνεται ακόμα και με το Google. Τελικά βέβαια μετά από την επιμονή του Google η κυβέρνηση ε, υποχώρησε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιου είδους παρέμβαση ε, στην προσπάθεια κάποιων ανθρώπων απλώς να ε, πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και που δεν θέλουν να συνεργαστούν με την κινέζικη κυβέρνηση ή δεν θέλουν να καταδώσουν ε, οποιουσδήποτε ε, ε, όποιους πολίτες της Κινέζικης Δημοκρατίας δεν θέλουν να εκφράσουν μια αντίθετη άποψη. Πράγμα που συνέβη και με τον κύριο Λιουξιαμπάο. Ε, εδώ πριν από 20 χρόνια γνωρίζουμε τι συνέβη. Ε, αυτό, αυτά τα ε, τραγικά γενέθλια θα πρέπει να τα θυμηθούμε. Αλλά πραγματικά δεν προσέξαμε όπως έπρεπε το τι συνέβη πριν από 20 χρόνια. Ας το κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Στάνοκ. Για άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Στάνο, και εδώ πέρα συζητάμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων στην Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το θετικό καθεστώ των κομμουνιστών του Πεκίνου είναι αποφασισμένοι να καταστήλουν πάσα φωνή διαφωνία. Όμω, εμεί δεν θα πρέπει να διστάζουμε εδώ στο κοινοβούλιο να τα καταγγείλουμε. Και αυτό διότι αυτό είναι υποχρέωσή μα. Είναι ε, χρέο μα προ ε, του, του, του, ε, ε, του ε, μάρτυρε αυτού όπω ο Λιού Μπάου. Ε, έχουν εφημωθεί και ε, αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Και επίσης ε, Χουτσία που κέρδισε το βραβείο Ζαχάροφ ε, καταδεικνύει ότι μας ενδιαφέρει το θέμα των δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Κίνα είναι τεράστια, ε, είναι πάρα πολύ ισχυρή στρατιωτικά, οικονομικά, οπότε θα πρέπει εμείς να δούμε πώς θα υπάρχει κάποια εταιρική σχέση ε, στη βάση της ισότητας, ε, του σεβασμού, της ασφάλειας, να δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε όμως και κράτος δικαίου και δημοκρατικές αρχές κοινές. Ελπίζουμε και κάποια στιγμή όλα αυτά τα ιδιώδη τα είναι ξένα προς την Ασία ελπίζουμε κάποια στιγμή όλα αυτά να ισχύσουν και στην ε, Κίνα. Να, ε, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ινδία, τεράστια χώρα, τι γίνεται στην Ταϊβάν. Εκεί υπάρχει ελεύθερη κοινωνία, οπότε μήπως και αυτοί μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις αξίες και στην Κίνα. Ευχαριστούμε κύριε Τάνακλε και τώρα για 1,5 λεπτό έχει το λόγο η κυρία Χαούταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό εδώ στην περίπτωση Ζιαμπάου είναι πως ε, βρέθηκαν και αυτοί οι 10.000 να τον υποστηρίξουν δημόσια και εγώ νομίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό ναι. Κοινοβούλιο πρέπει πραγματικά να σημειώσει το θάρρος αυτών των ανθρώπων και να τους ευχαριστήσει. Ταυτόχρονα πρέπει να θυμόμαστε πως η Κίνα υποσχέθηκε να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέλει να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και λέει πως θα δεσμευτεί για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα υποστηρίξει ε, τυχόν τέτοια αιτήματα. Αυτά έχει υποσχεθεί στον ΟΗΕ και πρέπει να τα θυμόμαστε. Επίσης το ψήφισμα αναφέρει τον ε, διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Όσο αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε, το αποτέλεσμα είναι πως ε, ο διάλογος αυτός δεν έχει ωφελήσει και πολύ. Μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βελτιώσουμε τη δική μας στρατηγική για να αντιληφθεί η Κίνα πως οι δεσμεύσεις της ε, στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που αφορά και εμάς και αυτούς και σε, εξαρτάται η συνεργασία μας από αυτό. Μπορούμε να ρωτηθούμε γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο κατακαιρματισμένη και τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την Κίνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια νέα στρατηγική με την Κίνα. Ευχαριστώ. Περνάμε στους ομιλητές εκ των πολιτικών ομάδων. Πρώτο, ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι λέξεις ε, δεν πρέπει να θεωρούνται ε, εγκλήματα. Αυτό είπε ο Λιού στο πολιτικό του μανιφέστο, το οποίο υπογράφηκε και από 10.000 άλλους ε, Κινέζους ο Λιού Τσαομπό για την, για την τόλμη του να μιλήσει ελεύθερα καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης. Γνωρίζουμε τη στάση της κινέζικης κυβερνήσεως κατά των ακτιβιστών των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων ε, ε, Ξέρουμε ότι ο κύριος υποκινητής ε, των γεγονότων της πλατείας Τιανανμέν και αυτός καταδικάστηκε ε, σε 9 χρόνια ε, φυλάκισης. Πιστεύουμε ότι, όπως και η κυρία Χαουτάλα είπε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας 29 Δεκεμβρίου του 2009 εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωση σχετικά με την εκτέλεση του Ακμάλ Σεϊχ ε, ε, και ότι βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε έναν ευρύτερο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό ο κύριος Μπαλσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μια νέα συμφωνία πλαίσιο με την Κίνα. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμο για ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με τη χώρα εκείνη. σημαντικέ αυτέ οι σχέσει. Όμω δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε πριν εξασφαλίσουμε σεβασμό ανθρωπινών δικαιωμάτων και κράτου δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναβαθμίσει τον διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη χώρα αυτή που ξεκίνησε το 2000. Και μέχρι στιγμή είναι ατελέσφορο και θα πρέπει ο υψηλό εκπρόσωπο να εξασφαλίσει συντονισμένες προσπάθειες και αποτελεσματικές προς εκείνη την κατεύθυνση για το ώστε να είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά να είναι το θεμέλιο για την πολιτική που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπατσίτης λέει ο Πρόεδρος και τώρα για ένα 1,5 λεπτό έχει κύριε Τρίπελ το λόγο. όταν πήρε του ολυμπιακού σου Κίνες, ε, τους Ολυμπιακούς Αγώνε με συγχωρείτε, έλβιζα και εγώ πως θα βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά κατά τη διάρκεια και μετά της Ολυμπιάδας διαπιστώσαμε πως είχαμε επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τώρα βλέπουμε, μετά την περίπτωση Λιού Ζαμπάο και την απαγόρευση ενός κόμματος ομοφιλοφίλων, πως φαίνεται πως περνάει μια εποχή των πάγων όσοι είναι πολιτικοί αντιφρονούντες και ομοφιλόφιλοι στην Κίνα. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε την απελευθέρωση του Λιου Ζαμπάου και να πούμε στην Κίνα πως εάν θέλει να αποτελέσει συνομιλητή της διεθνής κοινότητα, πως πρέπει να σταματήσει αυτά τα ιστερικά μέτρα λογοκρισίας και παρακολούθησης και ιδίως στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το πολιτικό φίλτρο του διαδικτύου είναι πλέον θεμελιώδες δικαίωμα η ελευθερία έκφρασης που πρέπει να την υπερασπιστούμε παντού. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα ίδια παντού, είτε εδώ, στη ΣΥΠΑ, στο Σουδάν ή στην Κίνα. Γι' αυτό πρέπει η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας να το συνηθίσει αν θέλει να παίξει έναν άλλον ρόλο και θεωρώ πως εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να το θέσουμε αυτό και στις συναντήσεις κορυφής. Ακριβώς γιατί χρειαζόμαστε συνεργασία και για την πολιτική του περιβάλλοντος, του κλίματος και τη χρηματοδότηση και τις χρηματαγορές. Πρέπει λοιπόν επιγόντως να αλλάξουν την πολιτική τους. Ευχαριστώ κυρία Τρούπελ. Για ένα λεπτό, κύριε Φοντάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, της Κίνας ε, αφορούν την αναγκαστική εργασία. Ε, αυτό το είδος σύγχρονης σκλαβιάς νομίζω ότι αφορά άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είμαστε βέβαιοι ότι πολλά από τα εμπορεύματα τα οποία προέρχονται από την Κίνα και έρχονται μέχρι τις χώρες μας οπωσδήποτε προέρχονται από την εργασία αυτών των ανθρώπων. Η Ευρώπη ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, πάρει μέτρα τα, ε, όσον αφορά τον αποκλεισμό εισαγωγής για εμπορεύματα τα οποία εξ ολοκλήρου ή εν μέρη έχουν παραχθεί σε αυτά τα κέντρα υποχρεωτικής εργασίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε όλα τα, όλα τα εμπορεύματα τα οποία μπαίνουν στην Ευρώπη να είναι ιχνηλάσιμα και επίσης να διέπονται από τις ίδιες αρχές και περιορισμούς ε, που αφορούν όλα τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξουν νόμοι και κανόνες ε, τους οποίους όμως θα σέβονται όλοι. Νομίζω ότι μονάχα απαγορεύοντας απλήρως την εισαγωγή προϊόντων τα οποία εν μέρη ή εξ ολοκλήρου έχουν κατασκευαστεί σε αυτά ε, τα κέντρα ε, αναγκαστικής εργασίας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ορθά το ρόλο μας σαν προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριος Μακμίλαν Σκότ. Είμαι, έχω την ε, τιμή να είμαι αντιπρόεδρος ε, ε, του Κοινοβουλίου για στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλάμε για τα θέματα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι στην ιστοσελίδα μου αναφέρω πάρα πολλά στοιχεία όσον αφορά την τελευταία μου τελευταία συνάντηση που είχα με αντιφρονούντες οι οποίοι είναι φυλακισμένοι ευτυχισμένοι. Ε, και βεβαίως ε, πρέπει να ε, αναφερθούμε ιδιαιτέρως και στην περίπτωση του Αχμάλ Σέλκ, ο οποίος εξαφανίστηκε ε, συγγνώμη, το, η περίπτωση του Ζάου Ζιζέγκ, ο οποίο ήταν χριστιανός ακτιβιστής και ο οποίος ε, ε όντας για τον Νόμπελ Ειρήνη, έχει εξαφανιστεί. Ε, γνωρίζουμε επίσης ε, ότι ο λόγος των ακτιβιστών πλέον γίνεται γνωστό σε ολόκληρη την Κίνα θα πρέπει να σιγουρευτούμε για την τύχη του Ζάο Ζιζέγκ και αν είναι φυλακισμένο να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να τον ελευθερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακμίλαν Σκότ. Θα δώσω το λόγο μονάχα σε δύο αγορητέ στην διάρκεια τη διαδικασία ε, Catch the Eye γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είναι 12 παρα 10, πρέπει να ψηφίσουμε στι 12 και έχουμε ακόμα ένα θέμα. Η κυρία Κρόα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχτούμε το ότι η οικονομική πολιτική έχει προτεραιότητα όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα ε, και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακολουθώ τις εξελίξεις σχέση με το Google και το, αυτή τη θεραλία κίνηση σταματήσει συνεργασία με την κυβέρνηση ε, για λόγους της λογοκρισίας που επιβλήθηκε. για τον ε, Τσαμπάου. Πάρα πολύ σωστά τα είπαν οι συνάδελφοι. Και θεωρούμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θίξει το ζήτημα αυτό στη συνάντηση κορυφή που θα γίνει. Άρα θα πρέπει αυτά να περάσουν από τι διαπραγματεύσει με την Κίνα και ε, να ξεκαθαριστεί ότι είναι λέντε τι οικονομικέ σχέσει με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Μάισλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε για το ποια είναι η σωστή παραλλαγή για να ασκήσουμε πίεση στην Κίνα γιατί εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα από την Κίνα. Γι' αυτό είπε η κυρία Ντεκάιζερ πως απέσυρε η ομάδα της στην υπογραφή της. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος γιατί ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον γράψει εγγράψει την Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, ευχαρίστω να την υποστηρίξουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο ο Λίου Ζιαμπάο, είναι και ο Γκάο ο οποίο εξαφανίστηκε και ακούμε υποτίθεται πως αυτοκτόνησε, αλλά δεν ξέρω, μάλλον με άλλον τρόπο πέθανε. Και είδαμε τι έγινε και στους ε, Ολυμπιακούς ε, αγώνες και γνωρίζει όποιο έχει επαφές με την Κίνα τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε δεν πρέπει, δεν είναι ο σωστός τρόπος πάντως τα κατεπήγοντα. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σαφώς την ανησυχία της για την δυσανάλογη ποινή του Λίου Ψιαμπάου 11 έτη δηλαδή φυλάκιση για τον ρόλο του επειδή συνέταξε τη χάρτα 08 ένα σχέδιο δηλαδή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταρρυθμίσεις στην Κίνα και για τη δημοσίευση κάποιων δοκιμίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ίντερνετ. Κύριε Πρόεδρε, εμείς αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ελευθερία έκφρασης και σκέψεις θεμέλια του δημοκρατικού μας συστήματος. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου είναι τελείως ασύμβατη με την ελευθερία έκφρασης και αντιβαίνει πολλές διεθνείς συνθήκες, οποίες έχει συνυπογράψει και η Κίνα. Επίσης, είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων του γενετήσιου προσανατολισμού, όπως ανέφερε και η κυρία Τρούπελ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποπειράθηκε να παρατηρήσει την δίκη και λοιπόν για το ότι εκδιώχθηκαν από την αίθουσα του δικαστηρίου παρατηρητές μας. Οι λεπτομέρειες που παρόλα αυτά μάθαμε για την δίκη δείχνουν σαφώς πως ο κύριος Λιού δεν είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπεράσπισή του και δεν είχε δίκαιη δίκη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να καλεί την κινέζικη κυβέρνηση να απελευθερώσει ανεφόρον τον κύριο Λιού και να δώσει τέρμα στην παρενόχληση και κράτηση των λοιπόν ατόμων που είχαν υπογράψει τη χάρτα αυτή. Γενικά η στάση μας σε σχέση με την Κίνα είναι μια στάση επικοδομητικής επαφής στο πλαίσιο της στρατηγικής μας σχέσης. Σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν καλωσορίσαμε την πρόοδο της Κίνας όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα όπως και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρές ανησυχίες ε, όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τις πρόσφατες εξελίξεις όπως αυτές που ανέφεραν οι βουλευτές στο πρόσφατο αυτό ψήφισμα. Οι ανησυχίες μας αυτές μεταφέρονται στις τακτικές μας επαφές και ιδιαίτερα στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις κινέζικες αρχές. Την τελευταία φορά, όπως ξέρετε, συναντηθήκαμε στις 20 Νοεμβρίου στο Πεκίνο. Η σχέση μας είναι τόσο ισχυρή ώστε μπορούμε να συζητούμε ειλικρινά αυτά τα, ειλικρινώς αυτά τα ζητήματα. Στο Αντζίνγκ, πέρυσι στην 10η Σύνοδο Κορυφής, θίξαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις συζητήσεις και στην συνέντευξη τύπου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βερτιά, η κυρία Κόρχολα ανέφεραν τις επιθέσεις κατά του Google. Η Κομισιόν θεωρεί πως αυτή είναι άλλη μία ανησυχητική εξέλιξη στο πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης στην Κίνα. Προφανώς παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν διαβουλεύσεις που συνεχίζονται μεταξύ της εταιρείας και των κινέζικων αρχών και θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και όταν θίγονται ευρωπαϊκές εταιρείες. Να σας διαβεβαιώσω κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, πώς θα συνεχίσουμε να φύγουμε αυτά τα ζητήματα και να το θέτουμε στο υψηλότερο επίπεδο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Να υπενθυμίζουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που περιέχονται στο Σύνταγμα της Κίνας αξιότυποι βουλευτές όλοι έχουμε τον κοινό στόχο μιας πιο ανοιχτή διάφανης Κίνας που θα τηρεί τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα συνεργάζεται μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες ευρωκλήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην εξέλιξη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Κύριε Πρόεδρε, Μία αντίδραση στο ερώτημα της κυρίας Ντεκάιζερ που μίλησε για την εκτέλεση του Βρετανού πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε ανεπιφύλακτα την εκτέλεση του Αχμαλσαϊ. Λυπούμεθα επίσης για το ότι η Κίνα δεν άκουσε τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός κράτους μέλους για τη φανατική ποινή του Ιουσάη για, και για την αναβολή εκτέλεσής της. Ο πρώτος. ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όμως, ακόμα, ακόμα λέγω, απομείνει ένα σημείο στη μερισσία διάταξη. Παρακαλώ καθίστε. Καθίστε και κάντε ησυχία. Θα συζητήσουμε τώρα το ψήφισμα σχετικά με τις Φιλιππίνες. Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια θλιβερή συνήθεια ε, αυτές ε, οι σειρές δολοφονιών